Αρχίζω με Αρχίζουμε τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν υπάρχουν. Υπάρχουν ενστάσεις. Όχι. Τα πρακτικά εγκρίνονται. Πρώτο θέμα, δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής,